Dear colleagues, we, we only have a limited time for votes. Um... Αδελφοί, λίγο χρόνο έχουμε. Μέχρι τις 12. Τότε συντομεύουμε. Okay, colleagues, settle down. Thank you. So we have the adoption of the agenda and if there are... Λοιπόν, καθίστε, εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ωραία, ευχαριστώ. Περνάμε κατευθείαν στο μόνο θέμα, ψηφοφορία για την θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα μετά την ψηφοφορία που έγινε χτες στην Επιτροπή στις 12 η ώρα. Συμφωνήσαμε η ψηφοφορία να γίνει σήμερα. Θα σας εξηγήσω λίγο την διαδικασία. Λοιπόν, η διαδικασία που συμφώνησαν σήμερα οι συντονιστές είναι η εξής. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού 2017-1939 ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου θα οριστεί Ευρωπαίος Αγγελέας για μία μία ανανεώσιμη θητεία 7 ετών. Εντάξει, ξέρω ότι πρέπει να οργανωθείτε για την ψηφοφορία, αλλά λίγο ήσυχα. Ακούστε όμως. Η οργάνωση τη ψηφοφορία είναι ω εξή. Όπω ξέρετε, στην επιστολή τη 21η Φεβρουαρίου, ο πρόεδρο Ταγιάννη ζήτησε μια κατάταξη των υποψηφίων. Στη σημερινή συνεδρίαση των συντονιστών αποφασίσαμε να γίνει μια ψηφοφορία ε, σε κάλπη μυστική με χάρτινα ψηφοδέλτια και έχετε νομίζω σας μοιράζουν τα ψηφοδέλτια Καθώς ε, δεν μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, θα ψηφίσουμε με κάλπη και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία είναι μυστική σύμφωνα με το άρθρο 180α και 181 του κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 180α εδάφιο 4 μεταξύ 2 ε, και 8 ε, βουλευτές, ένας αριθμός των ταξίδιων και 8 βουλευτών που θα επιλεγούν ε, με κλήρο, θα αποτελέσουν τους ψηφολέκτες. Να προτείνω τρεις λοιπόν. θέλω τρεις εθελοντές. Έχω ήδη την κυρία Σατζεντίνη και την κυρία Μέτσολα που έχουν συμφωνήσει. Κυρία Μακοβέη, θέλετε να είστε ψηφολέκτης. Όλοι θέλουν να είναι. Εγώ νόμιζα ότι δεν θα ήθελε κανείς. Πώς να γίνει τώρα χωρίς ε, να κοιτάξω. You put your hand up first. Η κυρία Μακοβέη σήκωσε το χέρι πρώτη, η κυρία Γκραπίνη δεύτερη. Τέσσερις να έχουμε. Μακοβέη, Γκραπίνη, Σαρτζεντίνη και Μετσόλα, οι τέσσερις κυρίες. Καλή τύχη. Λοιπόν, ακούστε με να υπενθυμίσω τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά Ζαν Φρανσουά Μπονέρτ, ε, Λαουρα Κοντρούτα Κεβέση και Αντρές Ρίτερ. Τα ψηφοδέλτια με τα ονόματά τους ε, σας μοιράζονται ήδη από τους κλητήρες. Όταν θα ψηφίσετε, μπορείτε να ψηφίσετε μόνο έναν υποψήφιο. Με σταυρό. Εντάξει, καθένα που μα βάλτε ένα σταυρό να τελειώνουμε. Λοιπόν, αν ε, ψηφίσετε, αν σταυρώσετε πάνω από έναν, ε, θα είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια πάνω από ένα όνομα θα είναι άκυρα, δεν θα ληφθούν υπόψη. Οπότε, επιλέξτε ένα όνομα και βάλτε το στην κάλπη θα ε, φωνάξω τα ονόματα των συναδέλφων για να έρθουν να ψηφίσουν. Και μετά θα επιστρέφετε στο εδρανό ή μπορείτε να φύγετε, αν θέλετε. Λοιπόν, αυτό είναι νομίζω ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να γίνει η ψηφοφορία. Επίσης, να πω το εξή. Μόνο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τη Επιτροπή μπορούν να ψηφίσουν εξαίρεση μπορεί να γίνει για πληρωματικά που δεν είναι μέλη της ΛΥΜΠΕ μόνο εάν το όνομα τους έχει γνωστοποιηθεί στο Προεδρείο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 200. Έχουμε ελέγξει τον κατάλογο λοιπόν, οπότε θα ε, φωνάζω και τα ονόματα για να υπάρχει διαφάνεια. Λοιπόν, θα ανακοινώσω τα αποτελέσματα όταν ε, μετρηθούν τα ψηφοδέλτια και ξεκινάω Λέει εδώ πέρα να ξεκινήσουμε με αλφαβητική σειρά, ξεκινώντας από το α, ούτε αυτό δεν με εμπιστεύεται να καταλάβω η γραμματεία. Λοιπόν, ξεκινάει η ψηφοφορία. Ε, έχετε κάποια ερώτηση, κάποια... κάτι να πείτε πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Μια στιγμή μόνο γιατί υπάρχει μια αλλαγή στον κατάλογο εδώ οι ε, ψηφολέκτες θα ψηφίσουν τελευταίες. Και κύριε Σαρτζεντίνη σας παρακαλώ τώρα πηγαίνετε εκεί στην κάλπη. Λοιπόν, διάλειμμα ενός λεπτού. Just increase the tension.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 Okay, colleagues, I'm now going to announce... Λοιπόν, συνάδελφοι, τώρα θα να πω τα ονόματα με αλφαβητική σειρά. Με αλφαβητική σειρά είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, όχι τα αναπληρωματικά. Λοιπόν, ο κύριος Αντάμοφ, τον οποίον αντικαθιστά ο κύριος Μπουσόελ. Is he here? Είναι εδώ. πραγματικά δραματικές οι στιγμές που ζούμε. Μαρτίνα Άντερσον. Is Martina here? Είναι εδώ η κυρία Άντερσον. Όχι. Μπάτεν, όχι. Μπέκερ. δόξα τω Θεώ. Παρόν. Η στιγμή έφτασε. Κυρία Μπένοβα την αντικαθιστά. Κύριος Πόπα. Then we have uh, Malin Bjork. Bjork. Η Μάλιν είναι εδώ. Okay. Mikael. Ωραία, Μίκα Αλμπόνη. And then Katerina Chinichi. And substituting for Daniel Do τον Ντανιέλ Ντάλτον τον αντικαθιστά ο κύριος Ντεμικέλη Desmacher Mr. Desmacher De Mesmacher for, for Mr. Dalton and then substituting και μετά την ε, Ρασίντα Αντατή, την αντικαστά ο κ. Λαβριλίου. Δίας Δεμέρα. Είναι εδώ, όχι. Φρανκ Έγγελ. Τον κύριο Δίας Δεμέρα δεν τον αντικαθιστά κάποιος. Μια στιγμή, μια στιγμή. Α, μάλιστα. Ε, η κυρία Γκρέσλη αντικαθιστά τον κύριο Ντεμέρα. My apologies. Uh, the replacement for Frank... Αντί του Φρανκ Έγγελ, ο κύριος Λέναρτ. και αντί της Κορνίλια Έρ στον κύριο Σομαρζέ. Um, the replacement for Tanya κυρία Γκραπίνη που αντικαθιστά την κυρία Φαγιόν. Ε, μπορείτε να ψηφίσετε, εντάξει, παρότι είστε ψηφολέκτρια. Λάουρα Φεράρα δεν είναι εδώ. Φίντ, ούτε εδώ. Και αυτό. Ο Ρώμεο Φράντ. Ε, Μούρεσαν αντί τη κυρία Κίνγκα Μούρεσαν Ο κύριος Μάμικιος πρωτοκαθιστά την Άννα Γκόμες, η Νατάλη Γκρισβέκ, Σιλβί Γκυγιόμ, Σιλβί Γκυγιόμ, Mr. Alaaho um, is replaced by... Κύριος Πάκετ, αντί του Αλάχο. I'll slow down. The tellers are asking me to slow. Α, τα πάω, τα λέω γρήγορα μου λένε οι ψηφολέκτε. Καλά, θα επιβραδύνω. Θα επιβραδύνω. Συγγνώμη συνάδελφοι. Γιατί πρέπει και να υπογράφουν οι συνάδελφοι, άρα θα προσπαθήσω να πηγαίνω πιο αργά. Monica Holmeyer, please. Η Μόνικα Χολμάιερ. Uh, Mr. Alahajo, yeah. And then Monica Holmeyer, then Bryce Hort.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 Όχι, δεν ανακοίνωσα, είπα. Α, είστε ψηφολέκτη. Μάλιστα. Εύα Ζολή. Είναι η Εύα εδώ. And Dietmar Koster, please. Τώρα ο Dietmar Koster, Kester. Oh, this is... Ms. we have no change. Sorry, just, just to check, um, are you voting... Για να το επαληθεύσω. Εσείς ψηφίστε αντίστοιχα σας μανόβερ. Γιατί δεν το είχαμε. Χουσμένοβα. Mr. Costa. Okay, replacing Barbara Kajiska is Miss, Mrs. Pitera. Pitera Dikatsiska. And Cecil Kienge, please. Okay Cecil Kienge. Mr. Mrs. Mrs. And replacing um, Mr. Lopez Aguilar. Αντί του κ. Λόπεθ Αγγιλάρ, κυρία Γκαρθία Πέρεθ. And uh, voting now, uh, and Monica McAvey can vote now. Monica. Η Μόνικα Μακοβέη μπορεί να ψηφίσει τώρα. Είναι έτσι πιο εύκολο. Δυστυχώς. Συγγνώμη. Βαλεάν. Αντί της Μπάρμπαρα Ματέρα. And Roberta Metzola, please. Η Ρομπέρτα Μετσόλα. Αντί του Λεμισέλ.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 της Αλσάντρα Μουσολίνη. Ο κύριος Μάνισαν. From the EPP. Το ΕΛΚ. Replacing Mrs. Mussolini. Can someone from the EPP help me with this? πάντων, να με βοηθήσει κάποιος από το ΕΛΚ. Ποιος αντικαθιστά την κυρία Μουσολίνη. Μάνε Σάου λέει κάτι στο Α, Μαρινέσκου λέει. Δεν το λέει έτσι εδώ στο χαρτί μου. Κύριε Μαρνέσκο, συγγνώμη. Thank you, Mr. Marinescu. Ευχαριστούμε κύριε Μαρινέσκου. Αντί του Ιωζεφ Νάρς, κύριο Σόλμπριχτ. Replacing Peter Niedermüller is... Αντί του Πέτρου Νίτερ Μίλλερ η Σιλβία Ιβόν Κάουφμαν. Yes. Um, replacing Ivari Padar is Mrs. Zoan. De Padar. Yeah, this one here. Uh, Mr. Payne, EFTD. Ο κύριος ε, Payne από το EFTD. Ο κύριος Πάβελ αντί της κυρίας Post. Judith Argentini, ο Τζαν Κάριο Σκότα, όχι δεν είναι εδώ, Μπέγκετ Ζίπελ, Πράνισλαβ Σκρίπεκ, δεν είναι εδώ, Τσάμπα Σόγκορ, replacing Mr. Stanishev is Mr. Ο κύριος and αντί για τον κύριο Πράνισλαβ and Helga Stevens Valdemar Tomaszewski. Ο κύριος Ουγκουρεάνου. Μποντίλ Βαλέρο. Η κυρία Βερζιάτ. Harald Filimski, Udo Voigt, η κυρία Τζούντιθ Καρτεντάλεν ε, στη θέση του κυρίου Βάιντεν Χόλτσα. Πίτερ Τζέζεκ αντί της κυρίας Βίξτρομ. Κριστίνα Βίνμπεργκ. Τόμας Τσετσόφσκι. ο κύριος Σέλστρα. και ένα μέλος που παραλείψαμε, η κυρία Σπινέλη αντί της κυρίας Μπιόρκ. Και Τέλος πρέπει να ψηφίσω κι εγώ. Έχουν ψηφίσει όλοι οι ψηφολέκτες. Ευχαριστώ τους ε, ψηφολέκτες, ευχαριστώ για την ε, βοήθεια. Οπότε τώρα θα σταματήσουμε τη συνειδρίαση για να μετρηθούν οι ψήφοι. Και στη συνέχεια είστε ευπρόσδεκτοι να επιστρέψετε, οπότε και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Θα αναρωτιέστε για πόση ώρα θα κρατήσει λίγο. Αν θέλετε να παραμείνετε στις θέσεις σας μπορείτε να το κάνετε ή θα μπορείτε να βγείτε έξω για ένα μικρό διαβηματάκι. Hey colleagues, um, if you're ready, we can announce the votes. Αν είστε έτοιμοι, μπορούμε να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Έχω την τιμή να ανακοινώσω ψήφισαν η, ψηφο, η ψηφοφορία ήταν 50. Μία λευκή ψήφος ο κύριος Πονέα 22, η κυρία Κοβέση 26 ψήφους και ο κύριος γήτα μία ψήφο. Και τώρα θα αποστείλω ψηφοφορείο, μία επιστολή στην, στον πρόεδρο της ε, διάσκεψης των πρόεδρων, που θα τον ενημερώσω για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε με τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, ούτω ώστε να καταλήξουμε συμφωνία σχετικά με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας στην ψηφοφορία. Η επόμενη συνάντησή μας είναι στις 11 Μαρτίου. Λήξη της συνεδρίαση.